της 24. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έληξε. Καληνύχτα σε όλους.